Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος κύριος Σβόμποντα έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού. Παρακαλώ κύριε Σβόμποντα. Κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να πω το εξή. Ε, αυτή τη στιγμή ε, που στερχόμαστε εμείς εδώ, ακριβώς αυτή τη στιγμή, αυτή την ίδια ώρα, γίνεται η κηδεία του κυρίου Κληρίδη. Δεν είναι από τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά ο κύριος ε, Κληρίδης αγωνίστηκε σκληρά για να γίνει η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να επενθυμίσω σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία αγωνίστηκε για την Κύπρο και αυτήν ακριβώς τη στιγμή γίνεται η ε, εξόδιους ακολουθία στην ε, Κύπρο. Πρόεδρος, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόγοντα. Έστειλα εκ μέρους του Κοινοβουλίου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώην πρόεδρου του κυρίου Κληρίδη. Και έχω την επιθυμία να μιλήσει επί της μηνύσης διάταξης ο συνάρχος κύριος Ουτζίας. Παρακαλώ κύριε Ουτζία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρόεδρε Σούλ. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς χθε τη νύχτα ένας κυκλώνας ε, έπληξε την περιοχή μου, τη Σαρδινία, τη δική μου πόλη μάλιστα, οδηγώντας σε δεκάδε θανάτους. Εγώ θεωρώ ότι ως μήνυμα αλληλεγγύα ε, πέραν της ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, το κοινοβούλιο αυτό θα μπορούσε και αυτό το ετούμε και εκ μέρου των συναδέλφων Μπαράτσο και Μπερλιγκουέρ αν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε ενό λεπτού σίγη για αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που υπήρξαν θύματα μιας φυσικής καταστροφής και που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη σκέψη μας και στις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο σας ζητάω ενός λεπτού σίγη κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ούτζιες, ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Θα επανέλθω γιατί έχω να κάνω και άλλες ε, παρεμφερείς ε, ανακοινώσεις. Η συνάδελφος κυρία Μπαρατσούζη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο συνάδελφος Ούτζας, η περιοχή μου η Σαρδενία επλήγει από τον κυκλώνα Κλεοπάτρα 18 νεκροί μέχρι στιγμής ε, σκεπάστηκαν καλλιέργειες ε, και χωριά με λάσπη και βροχή Ετούμε κύριε Πρόεδρε το λόγο για να εκφράσω την οδύνη και να κάνω μια έκκληση στο παρόν κοινοβούλιο ώστε να στραφεί στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δεσμευτούν πραγματικά για την ανοικοδόμηση για να θέσουν στη διάθεση τη περιοχή τα απαραίτητα κονδυλία μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφο κυρία Μπαρατσούζη. Ε, οι εκπρόσωποι των θεσμών είναι παρόντες ε, και φαντάζομαι ότι και το Συμβούλιο και η Επιτροπή έλαβαν υπόψη τους ε, την έκκλησή σας. Υποθέτω ο κύριος Μοργάντη θέλει να λάβει το λόγο. Φαντάζομαι ότι πρόκειται επί του ίδιου θέματος. Ναι, Πρόεδρε, απλά για να εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου στο πληθυσμό της Αρδενίας. Έναν πληθυσμό που λατρεύει τη γη του, που υπερασπίζεται τις παραδόσεις και την ταυτότητά του και γι' αυτό και εγώ, ομόφωνα με τους συναδέλφους, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη που θα μπορούσε να επιδείξει το Κοινοβούλιο, κάνοντας ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον πληθυσμό της Αρδενίας. Ευχαριστώ. Κύριε Τόμ, και εσεί επί του ιδίου θέματος, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να φυσικά πρέπει να επιδείξουμε λεγγύη στο λαό της Αρδινίας, αλλά να έχετε κατά νου ότι έχουμε μια παρόμοια περίπτωση όπως στις Φιλιππίνες που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και βλέπουμε για πρώτη φορά να συμβαίνουν τέτοια πράγματα λόγω της κλιματικής αλλαγής και ελπίζω λοιπόν ότι κάποια από εσά ε, θα ξανασκεφτείτε τις θέσεις ε, που έχετε λάβει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τούρνες. Ο κύριος ε, Καβαντά έχει δει το λόγο επί διαδικαστικού. Παρακαλώ κύριε Καβαντά. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Σύνοδο να δώσει σημασία και στην δολοφονία ενός Γαλλού δημοσιογράφου στο Μαλί πριν λίγες ημέρες. Ήταν ε, πραγματικά σοκ, τόσο μεγάλο σοκ που τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση να τηρήσει ένα λεπτό σιωπή, γιατί έχουμε δύο, δύο θύματα. Και φυσικά τα θύματα είναι και η ενημέρωση αλλά και η κοινή γνώμη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να επισημάνω ότι κανένα από αυτά τα θέματα που θίξετε δεν έχει σχέση με την ημερήσια διάταξη. Όσο δίκαιο και αν έχετε, ε, με παρεκάλεσαν οι συνάδελφοι από διάφορες χώρες οι οποίοι ασχολούνται με την κατάσταση στο Μαλί, αλλά κυρίως μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων με παρεκάλεσε να επαναλάβω αυτό το οποίο ε, έχω ήδη κάνει πριν ε, από μια εβδομάδα να συλληπούμε τους ε, δύο δημοσιογράφους που αναφέρθηκαν ε, τους εργαζόμενους του France International, του, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, να εκφράσουμε λοιπόν τα θερμά μας συλληπιτήρια. Και οι δύο δημοσιογράφοι ασκώντας ε, τα δημοσιογραφικά τους καθήκοντα και κάνοντας ρεπορτάζ για τη σύγκρουση, για τις έρηδες ε, στο Μαλί, κατέστησαν θύματα τρομοκρατών και δολοφονήθηκαν με αποτρόπαιο τρόπο. Οι δύο αυτοί δημοσιογράφοι κατ' ουσίαν εκπροσωπούν χιλιάδες δημοσιογράφων οι οποίοι πολύ συχνά γίνονται θύματα πολέμου, καταπίεσης και τρομοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν το ένα λεπτό σιγής ε, το οποίο θα τηρήσουμε για αυτούς τους δύο ανθρώπους αφορά βέβαια αυτούς τους δύο και αφορά τα αλληλέγγυα αισθήματά μας για τις οικογένειές τους, όμως κατ' ουσίαν αφορά ε, αυτό το λεπτό όλους εκείνους τους δημοσιογράφους οι οποίοι ασκώντας τα καθήκοντά τους διακυβεύουν ε, τη ζωή τους ε, και παράλληλα με το ένα λεπτό αυτός ε, θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα της καταστροφής στη Σαρδινία. Παρακαλώ να εγερθείτε. vielen dank! η αρμόδια επιτροπή υπέβαλε κείμενο με βάση το 216 ε, άρθρο 4. Η διόρθωση αυτή ε, γίνεται δεκτή. Εάν μέσα σε 24 ώρες ε, δεν ζητήσει κάτι διαφορετικό, ένας ικανός αριθμός μελών. Βλέπετε λοιπόν το θέμα αυτό που θα διατυπωθεί στα πρακτικά. Και ψηφίζουμε τώρα για την έκθεση Ντεχάνε και Κάλφιν σχετικά ε, με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι ονομαστική ψηφοφορία και είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψήφισαν